You need to press it. Πατήστε το κουμπί. To press the button, sir. No, Okay. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το λόγο για κάτι Το ήλεγξα με το Προεδρείο και ήμουν πρώτος. Δεν διαμαρτύρομαι γιατί δεν μου έδωσε το λόγο, αλλά γιατί έτσι όπως έγινε η διαδικασία, κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει όλοι στο catch και να μην γίνεται κατάχρηση της μπλε κάρτας. Να το ξέρω λοιπόν, να κάνω κι εγώ στην επόμενη συζήτηση δέκα ερωτήσεις με την μπλε κάρτα. Σας παρακαλώ πολύ, οργανώστε τη συζήτηση σωστά. stop Να σας εξηγήσω. Ήμουν παρούσα στη συζήτηση, την άκουσα με